Äh, Αρχίζει και πάλι η συνεδρίαση. Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας. Περνούμε τώρα στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας. Νέες υποψηφιότητες για τον τρίτο γύρο για το αξίωμα του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχω λάβει δυνάμει του κανονισμού. διατηρούνται οι υποψηφιότητες όπως είχαν και στο δεύτερο γύρο. Παρακαλώ τώρα τους κλητήρες να διανύμουν ψηφοδέλτια και φακέλους για την ψηφοφορία. Παρακαλώ τους ψηφοδέλτες να έρθουν στη θέση τους στις κάλπες. Οι ψηφοελέκτες παρακαλώ να λάβουν τις θέσεις τους. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπορείτε να μεταβείτε στις κάλπες να ψηφίσετε. Meine Damen und Herren. Κυρίες και κύριοι, ψήφισαν όλοι οι βουλευτέ. Ρωτώ ακόμη μια φορά. Υπάρχει κανείς που θέλει ακόμη να ψηφίσει, που δεν έχει ακόμα ψηφίσει. Τρίτη φορά. Θέλει κανείς ακόμη να ψηφίσει. Όχι. Πέραστες τις Κύριε Πρέτσελ, καταγράφετε στα πρακτικά η παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Σας ανακαλώ στην τάξη με τις συνέπειες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς. Διακόπτεται εδώ η συνεδρίαση. Με το κουδούνι θα κληθείτε να επιστρέψετε στην αίθουσα για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.